τα μέλη των Επιτροπών. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ζητεί ερμηνεία του άρθρου 191 σε σχέση με την Προεδρία ε, ε, μιας Επιτροπής. Μόνο τα τακτικά μέλη ε, βάσει του άρθρου 186 μιας Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν στο Προεδρείο αυτής αυτή η ερμηνεία θεωρείται εγκεκριμένη εάν μέχρι αύριο το πρωί, κυρίες και κύριοι, δεν διαφωνήσει μια πολιτική ομάδα ή 40 τουλάχιστον βουλευτές. Το κείμενο θα το βρείτε και στη διαδίκτυο στο Seance on Direct. Η συνάδελφος Χριστιάνα Μουσκαρτίνη μου διαβίβασε ότι στις 15 Οκτωβρίου προσχώρησε στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ερχόμαστε τώρα στη διάταξη των εργασιών.